δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα ε, τόσα εκατομμύρια πολίτε ζητούν νέα νομοθεσία. Εμεί ε, στην Ολομέλεια έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε αυτή τη νομοθεσία. Δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η γραπτή, ε, η γραπτή ερώτηση 50 των Μοντάλτο Βέλτα ε, Τάκουλα ε, σχετικά με το πρόγραμμα ΣΑΦ στα σχολεία. Έχει υπογραφεί επίσης από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών και σύμφωνα με το άρθρο 123 του εσωτερικού κανονισμού αποστέλλεται στους υπευθύνους και ε, εγγράφεται στα πρακτικά. Ε, ο κύριος Μπίνεφ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, Μάριο Μάουρο του ΕΛΚ, τον κύριο Μολτάρντο των Σοσιαλιστών, τον κύριο Τάκουλα των Φιλελευθέρων και βεβλέως το εκπρόσωπο των Ευρωπαίων Συντηρητικών οι οποίοι ε, υπέβαλαν μαζί μου την ε, δήλωση για το ε, να παίζουν σκάκι στα σχολεία πράγμα που δείχνει ότι δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και σύνορα πολιτικά ευχαριστώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ ο οποίος στήριξε αυτή την πρωτοβουλία και την έθεσε υπό την αιγίδα του να ευχαριστήσω την διοίκηση του Κοινοβουλίου για την εξαιρετική εργασία και όλους αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν την ε, δήλωση. Ε, πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τον Γιάννη ε, Γιώσοβιτ και τον Μίλα Σφέρ διότι δεν είναι μόνο κάτι καλό αλλά είναι κάτι καλό για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι στα, στα θεωρία είναι ο κύριος Ντανέοφ που είναι εδώ μαζί μας και στο τέλος θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο μετά την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπίνεφ. Κυρίες και κύριοι, πρωτού προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, ο συνάδελφος Λούτα Μπίσκι παρετήθη από πρόεδρος της Μπίσκη οπότε κύριε Μπίσκη καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εργασία σας σαν πρόεδρος της ΓΚΟΑ σας ευχαριστώ για την πολύ ανθρώπινη και συλλογική δράση σας και ήσασταν ένας πολύ πολύτιμο συνάδελφος θα παραμείνετε στο κοινοβούλιο αλλά εν ονόμη όλου του κοινοβουλίου σας ευχαριστώ για τη συνεργασία Βέβαια θέλουμε να συγχαρούμε και τη συνάδελφο Τσίμερ η οποία είναι η νέα πρόεδρος της πολιτικής ομάδας ε, και ε, τη συγχαίρουμε. Κυρία Τσίμερ, πρέπει να ομολογήσω όμως ότι τώρα ε, σας έδωσαν κίτρινο τριαντάφυλλο και όχι κόκκινο, οπότε θα μας εξηγήσετε γιατί. Σχετικά με το ε, εσωτερικό κανονισμό, οι φιλελεύθεροι ε, έχουν, ο κύριος Παπαστάμκος μάλλον έχει ζητήσει το λόγο. Προς εμάς και δημών προς το σώμα, όπως προταχθεί για ε, ευεξήγητους λόγους, η ψήφιση της έκθεσης του κυρίου, ε, συναδέλφου κυρίου Chris Davis. Σας ευχαριστώ.